καλωσορίσω στην αίθουσα τον μακαριότατο του Αρχιεπίσκοπο Χόρχε Ορτίγα, του συνοδεύοντε αυτών επισκόπου και ολόκληρη την αντιπροσωπεία τη επισκοπική διάσκεψη τη Πορτογαλίας. Είστε εδώ. Καλώ ήρθατε. Μακαριότατε, δράτω με τη ευκαιρία δράτω με της ευκαιρίες για να εκφράσω την αλληλεγγύη μας και τα συλληπιτήριά μας στο λαό της Πορτογαλίας και ειδικότερα στο λαό της Μαδέρα, που δοκιμάστηκαν τόσο σκληρά τις τελευταίες αυτές ημέρες. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας τους συνοδεύουν. Ο κύριος